Έχετε όλοι μαζί σας ε, την ταυτότητά σας. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά και επομένως θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως με το σημείο 8 της ημερησίας διατάξεως. Πρωτεϊνικό έλλειμμα στην ημερησία διάταξη. Ποια λύση σε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα. Η συγητής είναι ο Μάρτιν Χόσλινγκ. 132 τροπολογίες έχουν ε, υποβληθεί. Έχουν επίσης ε, ε, διαπραγματευτεί 11 τροπολογίες συμβιβασμού. Πιστεύουμε ότι ε, στο πέρας της ψηφοφορίας θα έχουμε ένα συγκερασμό των διαφορετικών απόψεων. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον Μάρτιν γιατί έχει ανακοινωθεί μια προφορική τροπολογία. Μάρτιν Χόισλινγκ. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, Βλέπετε ότι όταν υπάρχουν τόσες πολλές τροπολογίες σημαίνει πάντοτε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά επί του περιεχομένου και μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερες συμβιβαστικές τροπολογίες και ε, από τον ε, αριθμό των τροπολογιών βλέπετε ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σχεδόν ομόφωνα αλλά μέχρι το τέλος υπήρχαν και ε, προφορικές τροπολογίες οι οποίες στο τέλος αμφισβητήθηκαν αλλά οι συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες καταλήξαμε με τους οι συγητές θα έπρεπε να ισχύσουν για την Επιτροπή και ε, θα τις ψηφίσουμε έτσι. Έχω δύο σημεία που θέλω να αναφέρω. Καταρχήν ε, συζητήσαμε πολύ για τις ζωικές πρωτεΐνες όπου βρήκαμε ε, μία συμβιβαστική με την οποία θα μπορούσα να προχωρήσω και εδώ αναφέρομαι σχετικά με τη συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία όπου βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει επιτήρηση για τις πρωτεΐνες και γι' αυτό θεώρησα ότι πρέπει να υπάρξει μια τροπολογία. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να αποσιωπήσω τους, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς οι οποίοι κατά τη γνώμη μας ε, δεν πρέπει να περιληφθούν στην έκθεση διότι εμείς μιλάμε για την ευρωπαϊκή αγορά και όχι για ό,τι παρισφρεί από την πίσω πόρτα ε, με τις εισαγωγές της σόγιας και δεν θέλουμε να τις διευκολύνουμε ε, γι' αυτό και απορρίψαμε να κάνουμε συμβιβαστικές τροπολογίες επί του θέματος αυτού. Ε, έκανα μία έκκληση στους σκιώδεις εισηγητές ώστε αυτές οι τροπολογίες να αποσυρθούν. Ίσως σήμερα το πρωί κάτι θα συμβεί ακόμη, δεν έχω καμία ένδειξη προς το παρόν, αλλά ελπίζω ότι θα υπάρξει μια καλή ψηφοφορία στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Έχετε όλοι τον κατάλογο σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βουλευτές του ΕΛΚ, αλλά μονάχα 17 έχουν δικαίωμα ψήφου. Επομένως, επαλήθευση έτσι ώστε να γίνει ο αυτοέλεγχος. Ξεκινούμε λοιπόν την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής τροπολογίας 1. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία επί της συμβαστικής τροπολογίας 1. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και η καταδέμψη των ψήφων ε, είναι σωστή. Ποιο ζητάει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Δεν λειτουργήσε η κάρτα μου της ψηφοφορίας. Ναι, λαμβάνουμε υπόψη μα ε, λοιπόν, η γραμματεία θα λάβει υπόψη. Ενδεχομένως, εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί η κάρτα σας, ψηφίστε διανατάσσεω της χειρός. Ψηφοφορία επί του συμβιβασμού 2, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 95. 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ε, ναι, αλλά οι ομάδες θα πρέπει να δείξουν, να κάνουν μια ένδειξη ψήφου, λέει ο Πρόεδρος. Πέρα στις ψηφοφορίες επί του 95. Εγκρίνεται. Πέτα, βρε, πέτα. Αφού στα λέει. Εδώ έχουμε λοιπόν έτοιμα για προφορική ψηφοφορία. Πρέπει όμως ε, να σας ε, ρωτήσω εάν ε, είναι κανείς κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ψηφίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα. Α, όχι, μάλλον όχι. Πρώτα τι θα κάνουμε, θα ψηφίσουμε απευθεία, μπορούμε να ψηφίσουμε απευθεία. Ωραία, α ψηφίσουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία Ντόρφμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία Dorfman. Τώρα θα ψηφίσουμε την, την συμβαστική τροπολογία 3. Συμβιβασμός 3 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας επί του 3, το οποίο εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 99 Νικολέσκου, άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 99 Νικολέσκου. Πέρας Εγκρίνεται και η τροπολογία 99. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 100. Γκαρσία Πέρες. Άρχεται η ε, ψηφοφορία επί της τροπολογίας 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 100. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 101. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 101. Καλνιέται. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία 101. Ψηφίζουμε την τροπολογία 102. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 102. Εψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 102 εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβιβαστικής τροπολογίας 5. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106, Ρέιμερς και λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 106. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 106 εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 6. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 6. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 115. Λαβία. 115. Πέρας. Εγκρίνεται η 115. 117. Πρόκειται για μια προφορική τροπολογία. Συμφωνείτε όλοι με την προφορική τροπολογία 117 του κυρίου Λαβία. Να την ψηφίσουμε. Ωραία. Άρα άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 115. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7. Άρχεται η ψηφοφορία επί του συμβιβασμού 7. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία Ταμπάτζη 116, άρχεται η ψηφοφορία. Μάλλον όχι, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, συγγνώμη. Φτάνω, τώρα πάμε απευθεία στην, στο συμβιβασμό 8. Συμβιβασμό 8 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ε, εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία επί του συμβιβασμού 9. Συμβιβασμό 9. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Εψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 129. 129 Ρέιμερς και λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία επί της 129. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες ε, για την ε, τροπολογία 129 που απορρίπτεται. Τέλος, ε, τροπολογία 131 Νικουλέσκο, άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 131. Εψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται η 131. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Πέρας της πληροφορία. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 4. Ε, Σικιέρσκι. Ε, ψήφισαν όλοι επί της, 4, επί της ε, τροπολογίας 4. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Γκαρθία Πέρεθ. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Mm. 6. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Πέρας της ψηφοφορίας επί του 6. Επί 6. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 7 Λεφόλ. Εψήφισαν όλοι την τροπολογία 7. 7. Πέρας της ψηφοφορίας για την τροπολογία 7. Η οποία απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ψηφίζουμε την τροπολογία 8, άρχιδη ψηφοφορία. Uguale. Chiuso l'8. Πέρα στις 8. Η 8 απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 9. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 9, η οποία εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ψηφίζουμε. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η 10. 11. Ψηφίζουμε την τροπολογία 11. Πέραση. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 12. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Όχι, όχι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία ε, της τροπολογίας 13, Ρέιμερς και λοιπόν. Ολοκληρώθηκε. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία 13. Τροπολογία 14. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται η τροπολογία 14. Τροπολογία 15 καλνιέται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. 16. Δαντά. Ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 16. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται, 17. Νικουλέσκου. Ψηφίζουμε την τροπολογία 17. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται την τροπολογία 17. 18. Δαντά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 18. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 18. Ε, περνάμε τη 19, πηγαίνουμε στην 20. Τροπολογία 21, συγγνώμη. 21, 21. Τροπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία. Θεολογική σκέψη 21. Ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται η τροπολογία 21. 22. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 22. Πέρας. Εγκρίθηκε η τροπολογία 22. Πάμε τώρα στην τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 28. 28. Ψήφισαν όλοι για την τροπολογία 28. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία 28. Τροπολογία 29 Νταντάν. Άρχεται η ψηφοφορία από της τροπολογίας 29. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 29. Τροπολογία 30. Ψηφίζουμε την τροπολογία 30. Συμφωνούν. Εγκρίνεται λοιπόν. Όλοι συμφωνούν με την τροπολογία Λεφόλ. Τροπολογία 31. Ashworth. Άρχεται η ψηφοφορία από της τροπολογίας 31. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 31 εγκρίνεται. Votiamo sul 32 adesso. Ψηφίζουμε την τροπολογία 32 Νταντάν. Τροπολογία 32 Νταντάν. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Ψηφίζουμε την τροπολογία 34. Πέρας. Η τροπολογία 34 απορρίπτεται. 35. Ψηφίζουμε την τροπολογία 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η 35. 36. 36. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 36. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 36. Τροπολογία 37. Ψηφίσουμε για την τροπολογία 37. Πέρας. Η τροπολογία 37 απορρίπτεται. 38. Ψηφίζουμε λοιπόν επί της 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 38. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 38. 39. Άρχεται η ψηφοφορία από της τροπολογίας 39. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 39. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται η 40. 41. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 41. Εγκρίνεται η 41. 42 Μάγερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 42 απορρίπτεται. 43. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η 43. 44. Άρχεται η ψηφοφορία για την 44. Ψήφισαν όλοι. Πέρας η τροπολογία 44 απορρίπτεται. 45. Ψηφίζουμε η τροπολογία 45. 45 λοιπόν, η 45 εγκρίνεται. 46, ψηφίζουμε την τροπολογία 46. Λοιπόν. εψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται η τροπολογία 46. 47. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 48. Ψηφίζουμε για την 48. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 49. Θα ψηφίσουμε για την 49. Εγκρίνεται η 49. 50. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 50. Εγκρίνεται και η τροπολογία 50. 51. 51. Εγκρίνεται και η τροπολογία 51. 52, τα επίσης, ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται η 52 και περνάμε τώρα... Ναι, οι τροπολογίες Δαντάν ψηφίστηκαν. 55. 55. Πάλι Δαντάν. Σήμερα μόνο Δαντάν ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Εψήφισαν όλοι από τις 55. Εγκρίνεται. Σικέρσκι 56. εγκρίνεται. 57 λαβία. 57 λαβία. Εψήφισαν όλοι. Η 57 εγκρίνεται νομίζω, ε. Ναι, εγκρίνεται. 58, Γκοζές. Τροπολογία, λοιπόν, 58, πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 58. 59. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 59. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 59. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 60. Πέρας της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία 60. 61. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία 61 απορρίπτεται. 62. Άρχεται η ψηφοφορία από την τροπολογία 62. Πέρας. τροπολογία 62 εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 63, τροπολογία 63, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία εγκρίνεται η 63. Τώρα θα φτάσουμε στο συμβιβασμό 10. Οι τροπολογίες Λεφόρ και Νταντάν πάντα εγκρίνονται. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, λέει ο Πρόεδρος. Ε, συμβιβασμός 10. Συμβιβασμός 10 εγκρίνεται. Και φτάνουμε τώρα στην τροπολογία 71. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 71. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 72. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 72. 73. Τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Τροπολογία 73 εγκρίνεται. 76. Ταμπάζι Λεφόλ. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 76. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 76. Τροπολογία 77. Ψηφίζουμε την τροπολογία 77. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 77. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται και η τροπολογία 78 και φτάνουμε τώρα στο συμβιβασμό 11. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, δεν ακούν οι διερμηνείς. Ε, ε, ε, και, και ο Σιλβέστρης είναι υπέρ της τροπολογίας 78. λοιπόν, συμβιβασμός 11 εγκρίνεται ο συμβιβασμός 11. Α, δεν δηλώθηκε το πέρας της ψηφοφορίας. Ναι, τώρα είναι το πέρας της ψηφοφορίας και βλέπουμε ότι εγκρίνεται η τροπολογία, συμβαστική τροπολογία 11. Συμφωνείτε όλοι να δεχτούμε μία προφορική τροπολογία link επί της, ε, επί της 11. Ναι, επομένως ψηφίζουμε και την προφορική τροπολογία επί του συμβιβασμού 11. Εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τις τελευταίες ε, τροπολογίες. 84 γέγκλε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 84 γέγκλε. Πέρα της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 84 εγκρίνεται. Και τέλος, τροπολογία 85, άρχεται η ψηφοφορία επί της 8 πέρας εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε τις προτάσεις που μας έστειλε η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ψηφίσουμε μονάχα την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν επί της τροπολογίας 4 που προτείνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 4. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 5, πάντα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εγκρίνεται και η τροπολογία 5. Τροπολογία 6. Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πάντα. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6. Πέρας της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 6, η οποία εγκρίνεται. Και τροπολογία 9 της Επιτροπής Περιβάλλοντος πάντα. Άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Η τροπολογία 9 της Επιτροπής Περιβάλλοντος απορρίπτεται. Δεν μας είναι πολύ συμπαθής η Επιτροπή Περιβάλλοντος, λέει ο Πρόεδρος. Δεν θέλουμε την τροπολογία 9. Θα ψηφίσουμε τώρα στο σύνολο της εκθέσεως όπως έχει τροποποιηθεί. Επομένως έχουμε τελική ψηφοφορία στο θέμα του πρωτεϊνικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχεται η ψηφοφορία επί της εκθέσεως Μάρτιν Χάουσλινγκ. Εγκρίνεται. Ο κύριος Μποβέ ε, απέχει, αλλά δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας είπαμε, μπορούμε να συγχαρούμε τον συνάδελφο Μάρτιν Χάουσλινγκ. fate un punto della situazione. Bene, prendete una boccata d'ossigeno perché dobbiamo... Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα την έκθεση Παπαστάμκου. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, λέει ο Πρόεδρος, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. already to Papastankos? Yes. We have a lot of votes. Well, yes. yes. Passiamo ora alla votazione sul progetto di relazione di... Ψηφίζουμε τώρα ε, την ε, έκθεση ε, Γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνές Εμπόριο γεω, του κ. Παπαστάμκου. Έχουν υποβληθεί 127 τροπολογίες. Ο δε εισηγητής έχει υποβάλει τρεις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, Γιώργο, θέλεις να πάρεις το λόγο πριν αρχίσει η ψηφοφορία? Όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε άμεσα λοιπόν στην ψηφοφορία. Ξεκινούμε με την τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 18. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 19. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε συμβιβασμό 1. Άρχεται η ψηφοφορία του συμβιβασμού 1. Πέρας. Εγκρίνεται ο συμβιβασμός 1. Και περνάμε επομένω στην τροπολογία 25. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 25. Απορρίπτεται. Ναι, έπρεπε πρώτα να είχα δηλώσει, λέει ο πρόεδρος, το πέρας της ψηφοφορίας αλλά δεν πειράζει. Τροπολογία 27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της τροπολογίας απορρίπτεται η 27. Άρχεται η ψηφοφορία από της τροπολογίας 24. 24 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας η τροπολογία 24 απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 26. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Η τροπολογία 28 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 28. Πέρας της ψηφοφορίας επί της 28 απορρίπτεται η τροπολογία 28. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 29. Πέρας. Η τροπολογία 29 εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 30. Τροπολογία 30 λοιπόν πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία 30 απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Τροπολογία 31 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η 31 εγκρίνεται. Τροπολογία 37 ή μάλλον όχι, ζητώ συγγνώμη, τροπολογία 32. Τροπολογία Βοντσιεβόλσκι, ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 32. Εγκρίνεται η 32. Τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 37. Εγκρίνεται η 37. Τροπολογία 35 Νίκολσον. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 35. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας η τροπολογία 35 εγκρίνεται. Η 34 έχει καταπέσει, γιατί ψηφίστηκε η 37. 38, Μακγκίνες. Α, όχι, όχι, υπάρχει η, τροπολογία 36 του κύριου Ταραμπέλα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 36 του συναδέλφου Ταραμπέλα. 36. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Μα πώς το ψηφίσατε αυτή την τροπολογία 36, λέει ο πρόεδρος. Μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, 38. 38. Τροπολογία 38. Η τροπολογία 38 λοιπόν εγκρίνεται. 39 άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 39. Πέρας. Η 39 εγκρίνεται. Φτάνουμε στην τροπολογία 54. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 34. Σικιεύσκη. 54. Πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 42. 42 εγκρίνεται. 43. Τροπολογία 43, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε και την τροπολογία 45. πέρας της ε, ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας λέγω, απορρίπτεται η 45. Συμβιβασμός 2. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό 2. Εγκρίνεται ο συμβιβασμός 2. Τώρα θα ψηφίσουμε την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, ΙΝΤΑ. Άρχεται η ψηφοφορία επί της πρότασης ΙΝΤΑ. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. ναι, εδώ γράφει λέει ο Πρόεδρος ότι καταπίπτει αυτή η πρόταση εάν περάσει ο συμβιβασμό 2. Και από τη στιγμή που... Ε, όχι, δεν ψηφίζουμε γιατί εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε ο συμβιβασμός 2, επομένως αυτή η πρόταση από της παραγράφου 8 καταπίπτει. Και φτάνουμε επομένως στην τροπολογία 55. Ε, ε, ψηφίζουμε την τροπολογία 55. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 55. 55. Πρώτο τμήμα, ναι, είναι, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, είναι κατά τμήματα. Τροπολογία 55. Πέρας της, τροπολογίας, της ψηφοφορίας. Μου υπεδεικνύουν ότι ενδεχομένω υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στον κατάλογο ψηφοφορίας που έχετε εσεί μπροστά σα και τη γραμματεία που είναι πιο τελευταίο. Πρέπει να ακολουθείτε αυτά που σα λέω εγώ. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 57. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 57. Άρχεται η ψηφοφορία ε, επί της τροπολογίας 57 Ρόντουστ. Εψήφισαν όλοι επί της τροπολογίας 57. Πέρασε η ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 59 Γιάρ Τόρφμαν. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 59. πέρα της ψηφοφορίας από της τροπολογίας 59, η οποία απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 56, Άρχεται η ψηφοφορία από της τροπολογίας 56. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 56. Τροπολογία του εισηγητού, υπαριθμών 60. 60. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 60, πέρα στις ψηφοφορίες. Η τροπολογία 60 εγκρίνεται. Τροπολογία 61, ε, Σικέρσκι. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 61. Chiuso. Il voto. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται η τροπολογία 61. 62. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 62. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 62. 66. Ψηφίζουμε την τροπολογία 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, θα έλεγα εγώ. Ναι, απορρίπτεται. 63. τρία. Τροπολογία 63. Ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες επί της τροπολογίας 63. Απορρίπτεται. 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίες, Τροπολογία 64. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 67. Μάρκ Ταραμπελά. Συμφωνείτε όλοι με την τροπολογία αυτή. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία 67. 65. Ψηφίζουμε την τροπολογία 65 του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 65. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 68. 68. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 68 Βοτζεβόσκι. Εγκρίνεται η τροπολογία 68. Ψηφίζουμε τώρα την παράγραφο 13 γνωμοδότηση ίντα. Πρέπει να ψηφίσουμε αυτή τη φορά. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 13 έτσι όπως την έχει προτείνει η ίντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Επιτροπή ΙΝΤΑ πέρας. Απορρίπτεται για μία ψήφο. Τροπολογία 69 ρόντουστ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται η τροπολογία 69. Τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 Νίκολσον. Τροπολογία 71 Νίκολσον. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Παόλο Άλβες. 76. Τροπολογία 76. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 77 Dorfman, Γιάρ Dorfman. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας για την τροπολογία 77, η οποία απορρίπτεται. 78. Τροπολογία 78 Φοντάνα. 78. Τροπολογία 78. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81. Άρχεται η ψηφοφορία επί της ε, τροπολογίας 81. 1. Πέρας. Απορρίπτεται. 82. Άρχεται η ψηφοφορία της 82. 82. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 83. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 83. Εγκρίνεται. 84. Ψηφίζουμε την τροπολογία 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 86. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 86. Πέρας. Απορρίπτεται. 87. Άρχεται η ψηφοφορία από της τροπολογίας 87. Πέρας. Η τροπολογία 87 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση της ΙΝΤΑ, της Επιτροπής ΙΝΤΑ, επί της παραγράφου 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 88 του εισηγητού. Τροπολογία 88 του εισηγητού άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία 88 εγκρίνεται. Τροπολογία 89 άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 89. Γέγκλε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 92. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 93. Πέρας. Η τροπολογία 93 εγκρίνεται. 94. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 94. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 122. Herbert Dorfman. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τροπολογία 122 εγκρίνεται. Φτάνουμε τώρα ε, στην ψήφιση του συμβασμού 3. Άρχεται η ψηφοφορία επί του συμβασμού 3. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και πάμε απευθείας στην τροπολογία 105. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 105. Ο κύριος Ταραμπέλα, ε, ίσως είναι λεπτομέρεια πρόεδρε. Από τη στιγμή που η τροπολογία 101 δεν καλύπτεται από το συμβιβασμό, γιατί δεν το ψηφίζουμε και πάμε απευθείας στην τροπολογία 105, Πρόεδρος, η γραμματεία μου λέει ότι στην ουσία συμπεριλαμβάνεται στο συμβιβασμό. Επομένως ψηφίζουμε όντως την τροπολογία 105. Άρχεται η ψηφοφορία της τροπολογίας 105 Πόλσεν. Απορρίπτεται η 105. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 106 του εισηγητού. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 106, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την παράγραφο 5 που προτείνει η Επιτροπή Ίντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Εψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107 ακόμα ε, μία φορά του εισηγητού. Τροπολογία 107 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Η τροπολογία 107 μάλλον πέρασε της ψηφοφορίας και η τροπολογία 107 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την, την τροπολογία 108. Τροπολογία 108 έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Πέρα στις Η τροπολογία 108 απορρίπτεται. Έχουμε τώρα την τροπολογία 109, ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Τροπολογία 109, πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της 109. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Φτάνουμε στην τροπολογία 111 Νίκολσον. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 111. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 111. Τροπολογία 112. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 112. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται η 112. 113 Μάρκ Ταραμπελά, άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 113. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Τροπολογία 114. Άρχεται η ψηφοφορία της τροπολογίας 114. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Τροπολογία 115 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 115 πρώτο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορία. εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 115, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 116 Νίκολσον, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Έχουμε την ε, ε, πρόταση ίντα σαν προσθήκη. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμφωνούν όλοι από ό,τι βλέπω, άρα αφού κλείσω την ψηφοφορία λέω ότι εγκρίνεται και η πρόταση ίντα. Ακόμα μια τροπολογία του εισηγητού υπαριθμών 117 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 119. Άρχεται η ψηφοφορία της τροπολογίας 119. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία 119. Πρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση ίντα. Ε, προσθήκη και αυτή τη φορά. Ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 120. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 120. Συμφωνείτε. Ε, πέρας μάλλον της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται η 120. 121. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 121. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία 121. 123 του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 124, πολλοί συνυπογράφοντες. 124. Σίγουρα θα περάσει με τόσους συγγραφείς, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Παρατήρηση εκτός μικροφόνου δεν ακούνε διερμηνείς. «125 Ελίζαμπετ Γέγκλε, ε, τροπολογία 125 άρχεται η ψηφοφορία». Εγκρίνεται. Δηλαδή, ναι, πέρασε τη και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 126 Λορέντζο Φοντάνα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορίας απορρίπτεται. 127. Τροπολογία 127 του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε την παράγραφο 13 όπως την προτείνει η ε, Επιτροπή Ίντα. Πρέπει να ψηφίσουμε γι' αυτό. Επομένως άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Ε, ψήφισε, ψηφίσατε όλοι, κλείνουμε την ψηφοφορία, εγκρίνεται. Παράγραφος 14, πάντα πρόταση της ίντα. Ε, ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται η 14. Και μετά, παράγραφος 15, τελική πρόταση της Επιτροπής ΙΝΤΑ, ψηφίζουμε την παράγραφο 15 της πρότασης ΙΝΤΑ, περνάει, εγκρίνεται και έχουμε φτάσει τώρα στα εκτιμώντα. Ένα. Γρήγορα να πάμε, γρήγορα λέει ο Πρόεδρος. Ένα. Πέρα στις ε, ψηφοφορίες εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Τροπολογία 2. Εψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται η 5. 6. 6. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 8. Πέρας εγκρίνεται η τροπολογία 8. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Εψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι επί της τροπολογίας 10. Ναι, πέρας τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Τροπολογία 11 εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας η τροπολογία 9 εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας εγκρίνεται η τροπολογία 12. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία τη της τροπολογίας 16. Ψήφισαν όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 17. Ψηφίστε αυτή τη συλλογική τροπολογία. Εγκρίνεται. Τέλος. Έχουμε. Ναι, ναι, ξέχασα να ψηφίσω εγώ. Ναι, ναι. Αφαιρέθηκα, αφαιρέθηκα από τα τόσα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, να, θα, θα καταγραφεί η θετική μου ψήφος. Ναι, τώρα ψήφισα, τελείωσε. Τώρα έχουμε την ε, ψήφο επί των προτάσεων της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ε, Επιτροπή ΔΕΒΕ, παράγραφος 1, άρχεται η ψηφοφορία. Προτάσεις Επιτροπής Ανάπτυξης λοιπόν. 1. Παράγραφος 1. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. 2. Ψηφίζουμε την παράγραφο 2 των προτάσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. 2-2. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, ναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Εγκρίνεται πάντως. 3. Ψηφίζουμε την πρόταση, ε, την παράγραφο 3 της πρότασης Εγκρίνεται. Ε, το 6. Ψηφίζουμε την παράγραφο 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία από της παραγράφου 6. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίες από της παραγράφου 6. Απορρίπτεται. Επί της παραγράφου 7, ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της παραγράφου 7, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία επί του δεύτερου τμήματος του παραγράφου 7. Βλέπω ότι οι σοσιαλιστές ψηφίζουν έτσι λίγο διαφοροποιημένα. Τέλος πάντων. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την παράγραφο 8. Άρχεται η ψηφοφορία επί της ε, παραγράφου 8 της πρότασης. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα, θα ψηφίσουμε επί του συνόλου του ψηφίσματος, όπως έχει τροποποιηθεί, τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια Γιώργο Παπαστάμκο. Ακόμα μια αναπνοή για να περάσουμε και στα επόμενα.

Μια βασική πληροφορία. Λόγω του ότι υπάρχει αθρώα προσέλευση, σήμερα το απόγευμα στις 3 η, η ακρόαση θα γίνει στο ημικύκλιο, στην Ολομέλεια δηλαδή. Και θα έχουμε την αίθουσα της Ολομελίας για τη συνάντηση με όλους τους προσκεκλημένους. Και τώρα μια τελευταία προσπάθεια θα χρειαστεί να ψηφίσουμε την ε, έκθεση της κυρίας Γέγλε «Ο ρόλος των γυναικών στη Γεωργία και τις αγροτικές περιοχές» η συγγήτρια κυρία Γέγλε. Ε, έχουμε ε, ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών και κατάφερε η συγγήτρια να περιλάβει ε, τα θέματα σε 7 συμβιβαστικές τροπολογίες. Το λόγο έχει η συγγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όλους αλλά και τους χειώδης συγγητής και τους ε, βοηθούς ε, να τους ευχαριστήσω για την επικοδομητική συνεργασία. Δεν πίστευα ότι εκ των έξω θα υπήρχε τόσο ενδιαφέρον και καλή συνεργασία αλλά το βλέπουμε από τον πολύ ψηλό αριθμό των τροπολογιών και αυτό που καταφέραμε είναι να υπάρχει μία ακριβής ε, γραμμή στην έκθεση μετά από τη σημερινή ψηφοφορία όσον αφορά τις ε, ε, τις ε, θέσεις των συμβουλευτικών επιτροπών και θέλω να αναφερθώ σε ουσιαστικά τρία σημεία. Δηλαδή η δικιά μας σκοπιά από πλευράς της Επιτροπής Γεωργίας ε, αναφέρεται και στον οικονομικό αλλά και στον κοινωνικό ρόλο των γυναικών στις υπαίθρου και του χώρου της γεωργίας αλλά και το πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε διότι δεν θα πρέπει να υπάρχει μία δυσμενή μεταχείριση και διάκριση κατά των γυναικών και γι' αυτό προσπάθησα να ε, παρουσιάσω τις συμβαστικές τροπολογίες και θα τις συμπληρώσω με μια προφορική τροπολογία. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ είναι το θέμα της ενίσχυσης των μεταφορών στην υποδομή. Η υποδομή είναι αναγκαία εις τον αγροτικό χώρο αλλά οι μεταφορές πρέπει να συμπεριληφθούν εις τη συζήτηση για το μέλλον της γεωργίας και άρα δεν μπορούμε να προκαταλαμβάνουμε εδώ. Ε, γι' αυτό και ε, είδα ότι ε, χθες υπερψηφίστηκε μία έκθεση και μία τροπολογία σχετικά με την ενίσχυση της χρηματοδοτήσεως του δικτύου μεταφορών. Εγώ όμως δεν μπορώ να ζητήσω στον δεύτερο πυλώνα χρήματα για τις μεταφορές στη Γεωργία. Βλέπω ότι υπάρχουν, υπάρχει όμως μία τροπολογία στο σημείο 100, στην τροπολογία 131 και προφορικά θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, οι γεωργικές επιχειρήσεις. Η διατύπωση αυτή είναι πάρα πολύ σκληρή και θα μπορούσε να εξεταστεί εις ε, την ε, Εύχομαι... Ε, επικουρικότητα μεταξύ κρατών μελών. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη διατύπωση η οποία ε, να περιλαμβάνεται εις το ουσιαστικό κείμενο γι' αυτό και ζητάμε να στηρίξουμε την θέση των γυναικών κατά τρόπον ώστε ουσιαστικά αλλά και επαγγελματικά να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους εις την οικονομική ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει ε, μία ε, απόρριψη της τροπολογίας και να επανέλθουμε στο αρχικό κείμενο. Ε, κατόπιν αυτού προσβλέπω ή στην ψηφοφορία και ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους. Ευχαριστώ, είναι σαφές. Οπότε κατόπιν αυτού ξεκινάμε μέσα αμέσως στην τρο... τις ψηφοφορίες και ξεκινάμε με την πρώτη συμβιβαστική. Ξεκινά ψηφοφορία για την πρώτη συμβιβαστική. Λίγη. Η, η, η πρώτη συμβιβαστική υιοθετείται. Τροπολογία 39. Ξεκινά η ψηφοφορία για την 39. Λίγη. Η 39 περίφθη. 40. Ψηφίζουμε την τροπολογία 40, άρχεται η ψηφοφορία, λίγη, απερίφθη. 41, ξεκινά ψηφοφορία. Ε, ψηφίζουμε, λίγη ψηφοφορία, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 7 και ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 7, ξεκινά ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, λίγη ψηφοφορία και εγκρίνεται η συμβιβαστική 7. Τώρα ψηφίζουμε τη 42. 42 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, λίγη, η 42 απερίφθη. Ψηφίζουμε την 44. Ξεκινά ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 44. Λίγη. Απερίφθη αλλά δεν λειτουργεί το μηχάνημα του κυρίου Ντοντά. Τώρα ψηφίζουμε τη 46. Με συγχωρείτε 45 πρώτα. Πρώτα 45 ψηφίζουμε. λίγη. Απερίφθη. 46. Ξεκινά ψηφοφορία για τη 46. Ξεκινά. Λίγη. Απερίφθη. 47. Τροπολογία 47 ματέρα. Ξεκινά ψηφοφορία. Λίγη εγκρίθηκε. 48. Ψηφίζουμε τη 48. Ξεκινάει η ψηφοφορία στη 48. Λίγη. Απερίφθη. 50. Ψηφίζουμε την 50. Λίγη. Απερίφθη. 49. Ξεκινάει η ψηφοφορία 49. Λίγη. Εγκρίθηκε. 51. Τροπολογία 51. Ψηφίσατε. Κλείνει. Απερίφθη. 52. Ξεκινά. Κλείνει. Εγκρίθηκε. 53. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 53. Λίγη. Εγκρίθηκε. 54. Ξεκινά η ψηφοφορία για την 54. Λίγη 54. Εγκρίθηκε. 55. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 55. Εγκρίθηκε. Τώρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική 2. Ξεκινά η ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 2. Ψηφίζατε όλοι. Λίγοι. 63. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίθηκε. Τώρα ε, ψηφίζουμε τη συμβαστική 3. Ξεκινά ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη. Εγκρίθηκε. 72. Τροπολογία 72 ψηφίζεται τώρα. Με συγχωρείτε. Υπάρχει όμως και μία προφορική τροπολογία. Κάποιος αντιτίθεται, όχι. Οπότε εφόσον συμφωνούμε μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική Γκαρσία Περές. Ε, εγκρίθηκε. 74. Ξεκινά ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απερίφθη. 75 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Κλείνει. Ε, περίφθη 75. <coughs> Ψηφίζουμε την 76. Και η 76 έχει, είναι ψωροφορική, Αν κανείς δεν αντιθεί, αντιτίθεται ψηφίζουμε ε, λίγη ψηφοφορία εγκρίθηκε. 77. Ψηφίζετε την 77. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Αποτέλεσμα. Απερίφθη. 78. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφορία για την 78. Λίγη. Απερίφθη. 79. Δεκάστρο. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία του Προέδρου. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. 80. Υπάρχει ένας ο, ο οποίος όμως απήχε και θα τον βρω. Τροπολογία 80. Ψηφίζουμε την 80 ηλεκτρονικά. Λίγοι. Απερίφθη. 81. Τροπολογία 81. Ξεκινά. Ψηφίσατε. Λίγη. Εγκρίθηκε. 82. Ξεκινάει η ψηφορία για την 82. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Απορρίφθηκε. 83 σε δύο τμήματα. Πρώτο μέρος, ψηφίζουμε το πρώτο μέρος της 83. Κλείνει η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. Δεύτερο μέρος, δεύτερο μέρος της 83. Ψηφίσατε λίγοι. Απερίφθη. άλλη προφορική τροπολογία η 84 συμφωνείτε όλοι τότε ψηφίζουμε την 84 ξεκινά λίγη εγκρίθηκε 85 ξεκινά η ψηφοφορία για την 85 Νίκολσον λίγη η ψηφοφορία απερίφθη 86 Ξεκινά ψηφοφορία για την 86. Λίγη. Απερίφθη. 88. Ψηφίζουμε την 88. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβιβαστική 4. Ψηφίσατε, λίγοι, εγκρίθηκε. 97. Με συγχωρείτε. Έχετε δίκιο, πρέπει να ψηφίσουμε και την τροπολογία 89 που δεν ψηφίστηκε προηγουμένως, άρα ξεκινά ψηφοφορία για την 89. Ψηφίσατε όλη την 89, κλείνει η ψηφοφορία, εγκρίνεται. Τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε και την 90. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 90. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι εγκρίθηκε. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα και με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Εφόσον ψηφίσαμε τη συμβαστική 4, προχωρούμε στην 97 Reimers. Ποιος είναι υπέρ ε, ηλεκτρονικά, ψηφίσατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία, απερίφθη. 98. Ξεκινά ηλεκτρονικά, λίγη, απερίφθη. «99 τώρα» ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 99 η οποία εγκρίνεται. Έχουμε την ε, προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Η κυρία Λούλινγκ όμως ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είμαι η συγγήτρια αυτής της τροπολογίας και θα ήθελα να σας πω ότι... Όχι, όχι. Είμαστε ακόμη στην ε, προφορική τροπολογία, αλλά θέλω να σας επισημάνω την ε, κακή μετάφραση διότι δεν πρέπει να μιλάμε για πρεστασιόν maternal αλλά prestation de protection de maternité δηλαδή ε, για τις ε, υπηρεσίες για να προστατευθεί η μητρότητα δηλαδή ήθελα να αναφέρεται και για εκεί αναφέρεται και η τροπολογία μου περί τίνος πρόκειται για την προστασία της μητρότητος δηλαδή απλώς υπενθυμίζω τι ε, λέγεται εις ε, την οδηγία που αναφέρεται στους συζύγους που ασχολούνται με τη γεωργία. Ε, ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Γέγκελ να εξηγήσει στην συνάδελφο Λούλινγκ. Εγώ πιστεύω ότι το αρχικό κείμενο καλύπτει και την ανησυχία της κυρίας Λούλη διότι ε, αναφέρεται στην σχετική οδηγία και δεν μπορούμε ε, να επαναλαμβάνουμε σε κάθε παραπομπή το κείμενο της οδηγίας γιατί εδώ λέγεται σύμφωνα με την κυρία Λούλινγκ ότι πρέπει να υπάρχει επαρκή κάλυψη για τις συζύγους των γεωργών και για τις ε, γυναίκες για θέματα μητρότητος αλλά πιστεύω ότι καλύτερα θα το καλύψουμε με τη γενική διατύπωση παρά με τις λεπτομέρειες και γι' αυτό προτείνω να παραμείνουμε στην αρχική διατύπωση. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την κυρία Γέγλε αλλά πρέπει να ρωτήσω την κυρία Λούλινγκ αν συνεχίζει να διαφωνεί εκτός και αν συμφωνεί με την κυρία Γέγλε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να περιλάβουμε ακριβώς τη διατύπωση της οδηγίας διότι όσοι διαβάζουν αυτό το κείμενο της οδηγίας 2010-241 πρέπει να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και ε, αυτό θα ήθελα. Λοιπόν, συμφωνείς να ψηφίσουμε ε, όταν θα ψηφίσουμε την 100 να λάβουμε υπόψη τα σχόλια της κυρίας Λούλινγκ. Ωραία. Τώρα ψηφίζουμε την 100. Ψηφίσατε όλοι την 100, Λούλινγκ, ε, ε, εγκρίθηκε. 101. Όχι. 102. Άρκιν. Χάρκιν. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι την 102. Λίγοι. Απορρίπτεται. 103 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγοι. εγκρίθηκε. Δεύτερο μέρος της 103. Ψηφίζεται. Λίγη και εγκρίθηκε. Τώρα πάμε στην 106 Νίκολσον, ηλεκτρονική ψηφοφορία για τροπολογία 106. Κλείνει. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 5. Ξεκινά ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε. Εκατόν Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία στην 116. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 6 ξεκινά ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίθηκε. Εκατόν Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 121. Ψηφίσατε. Λίγη. Απερίφθη. Εκατόν εικοστρία. Τροπολογία 123 ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Λίγη. Απερίφθη. 124. Ξεκινά ηλεκτρονικά. Λίγη. Εγκρίθηκε. Όχι, με συγχωρείτε, απερίφθη. Σωστά το είχα δει στην αρχή, λέει ο πρόεδρος. 125. Ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη. εγκρίθηκε. 126. Ξεκινάει η για την 126. Λίγη. Απερίφθη. 127. Ξεκινώ την ψηφοφορία για την 127. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Εγκρίθηκε. 128. Έχουμε τώρα την 128. Ψηφίσατε όλοι την 128. Λίγοι. Απερίφθη. Προφορική τροπολογία πάντοτε της κυρίας Γκαρσία Περές. Κάποιος αντιτίθεται, όχι, ψηφίζεται ηλεκτρονικά η 129. Εγκρίθηκε. 130. Ξεκινά ηλεκτρονικά ψηφοφορία για την 130, λίγη, εγκρίθηκε. 131. Ξεκινά ηλεκτρονικά, λίγη, απερίφθη. 132. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Λίγη.

ξεκινά λίγη απερίφθη μάλλον αιτιολογική έκθεση 1 Γκαρσία Περές ξεκινά λίγη εγκρίθηκε εκτιμώντας ε, τροπολογία 2 απερίφθη εκτιμώντας 3 μάλλον ε, εκτιμώντας α3 τροπολογία λίγη εγκρίθηκε τροπολογία 4 ψηφίσατε απερίφθη. 6. Τροπολογία 6 για τα εκτιμώντας. Εγκρίθηκε. 7. Τροπολογία 7 για τα εκτιμώντας. Λίγη. Απερίφθη. 8. Ξεκινάμε την ε, ε, ψηφοφορία. Λίγη απερίφθη. 9. Τροπολογία 9. Ξεκινά ηλεκτρονικά. Λίγη εγκρίθηκε. Έχουμε άλλη μία προφορική τροπολογία της κυρίας Γέγκλε, της εισηγητρίας. Την ε, ψηφίζουμε. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, λίγη, εγκρίθηκε. 12. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 12. Λίγη εγκρίθηκε. 13. Ε, προφορική τροπολογία της Ντάντσλα. Αν κανείς δεν αντιτίθεται ψηφίζουμε. Ξεκινά η ψηφοφορία. Λίγη και ε, ε, ε, εγκρίθηκε. 16. 16 Μόσερ λίγη απερίφθη 18 ψηφίσατε όλοι λίγη 18 Εγκρίθηκε 19. Απερίφθη. 20. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 20. Ψηφίσατε όλοι. Απερίφθη. 21. Ψηφίζουμε την 21 τώρα. Ψηφίσατε όλοι την 21. Λίγη. Απερίφθη. 22. Ξεκινά ψηφοφορία για την 22. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη απερίφθη. 23. Μάλλον Μα, ε, συγχωρείτε 24 ξεκινά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 24 λίγη απερίφθη 26 σε δύο τμήματα για το πρώτο τμήμα ξεκινά ηλεκτρονικά ψηφοφορία Λίγη. Εγκρίθηκε. Δεύτερο μέρος της τροπολογίας 26 ξεκινά. Λίγη. Απερίφθη. 27. Τροπολογία 27. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη. Απερίφθη. 29. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 29. Ψηφίσατε όλοι. λίγη. εγκρίθηκε. 30. Ψηφίζουμε την τροπολογία 30. Ηλεκτρονικά. λίγη. Απερίφθη. Και τέλος η τροπολογία 31 σε δύο χωριστά τμήματα. Ξεκινά η ψηφοφορία για το πρώτο μέρος της 31 Λίγη. Εγκρίθηκε. Δεύτερο μέρος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απερίφθη το δεύτερο μέρος της 31 και τελική ψηφοφορία για την έκθεση Γέγκλε με τις ε, τροποποιήσεις που υπέστη. Ψηφίσατε όλοι, λίγοι. Εξαιρετικά συγχαίρουμε την ε, κυρία Γέγλε, μία από τις γιαγιάδες της ε, Γεωργίας και της Υπέθρου. Εγκρίθηκε η έκθεσή της. Ωραία, να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα. Να συνεχίσουμε λέω. Α, ένα λεπτό να κάνουμε stretching, λέει ο πρόεδρος. Prendiamo il lavoro e iniziamo con il punto 11 dell'ordine del Σημείο 11 Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Νορβηγία, όσον αφορά επιπλέον ε, συμφωνίε προτιμησιακέ. Πρόκειται για την έκθεση Richard Ashworth. Η πρόταση αυτή προτείνει αύξηση των ε, ε, διαπραγματεύσεων και τα, μάλλον τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων τα οποία συζητήθηκαν μεταξύ του Μαρτίου 2008 και μέχρι 8 ε, έχουν περαιτέρω και διεξοδικά συζητήσει στο θέμα σχετικά με εχορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, έτσι ώστε αφενός να απελευθερωθεί ε, περίπου το 60% των ε, γεωργικών ανταλλαγών μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για προϊόντα ε, ευαίσθητα όπως είναι το κρέας, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν δοθεί κάποιες ποσοστώσεις δασμολογικές καθώς επίσης και κάποιες μειώσεις. Όσον αφορά ε, κάποιες ειδικέ ε, διατάξεις, αυτές έχουν ε, προτεθεί και αφορούν τη διαχείριση των ποσοστώσεων σχετικά με το τυρί. Ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση, δίνοντας πρώτο το λόγο στο συντάκτη της νομοδότησης, Ρίτσαρντ Άσουερθ. Ρίτσαρντ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο, όπως πολύ σωστά είπατε. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου είναι η καθήλυνα αρμόδια για την έκθεση, αλλά η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για τα εμπορικά γεωργικά προϊόντα. Όπως ε, είπατε και νωρίτερα, με βάση τη συμφωνία η οποία εκπονήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φόρου, προβλέπεται η διμερής αναθεώρηση των ε, λεπτομεριών ε, της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας. Υπάρχει μια συμφωνία κυρίων για τους δεσμολογικούς ε, φραγμούς, προδευτική μείωσή τους δηλαδή. Και αυτό έγινε βάσει ανταλλαγής επιστολών. Τώρα, ε, με βάση τις ε, ισχύουσες προτάσεις ζητείται υπεραιτέρω απελευθέρωση των εμπορικών προτιμήσεων, πλήρης απελευθέρωση ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων και το 60% των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βασιλείου Νορβηγίας θα είναι πλέον εντελώς ελεύθερα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κανένας δασμός. Έχουν υπάρξει συμφωνίες και για άλλα πιο ευαίσθητα προϊόντα όπως είναι το κρέας, τα γαλακτοκομικά, ποροκυπευτικά, διακοσμητικά φυτά. Έχουν συμφωνηθεί ε, δασμολογικές ποσοστό σημειώσει των δασμών σε όλες τις περιπτώσεις και επίσης έχουν συνταχθεί δικές διατάξεις για το τυρί, όπου υπάρχει συμφωνία 7.200 τόνοι υπάρχει η συμφωνία να περιληφθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις. Απόλυα δοσμολογικών εσόδων, περίπου 4,96 εκατομμύρια. Αυτές είναι δημοσιονομικές επιπτώσεις και θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ε, η έκφραση των ευχαριστειών μου προς το προσωπικό της Επιτροπής μας που έκανε πολύ καλή δουλειά για την έκθεση αυτή. Και Αγαπητέ Πρόεδρε, θα ε, συστήσω στα μέλη της Επιτροπής να δώσουν θετική ε, γνωμοδότηση για την έκθεση. Ευχαριστώ, Ρίτσαρντ. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα. Σας πληροφορώ ότι... Ε, ναι, έχει ζητήσει ο κύριος Λαδία, ε, σας πληροφορώ ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 17η Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας εδώ θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου. Συγγνώμη, 27 Ιανουαρίου η κατάθεση των τροπολογιών 7 ε, Φεβρουαρίου. Να ακούσουμε τον κύριο Λαβία. Τζοβάνι, έχει το λόγο. Ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδα ότι στην πρόταση συμφωνίας με την Νορβηγία ε, υπάρχουν κάποια παραρτήματα ε, στα πλαίσια των οποίων έχουν, ε, γίνεται σαφή αναφορά στα προϊόντα. Και βλέπω διαρκώς αναφορά στα εσπεριδοειδή με εξαίρεση τα πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια δεν αναφέρονται σε καμία κατηγορία. Επομένως, θα είναι, ποιο θα είναι το καθεστώς για αυτά τα προϊόντα γιατί ξέρουμε ότι από, τις, τη νότια ε, Ιταλία οι εξαγωγές εσπεριδοειδών και βεβαίως και πορτοκαλιού είναι πολύ σημαντικά. Πολύ γρήγορα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να απαντήσει. Εδώ έχω σημειώσει ότι υπάρχουν τρεις εκπρόσωποι της Επιτροπής. Κλάρκ, Χίμοβα. Ποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ. Τζον Κλάρκ λέγομαι, μόλις ορίστηκα στη θέση του Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων για τον τομέα της Γεωργίας και ελπίζω να συνεργαστούμε πολύ καλά τους επόμενους μήνες για τα γεωργικά θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Άσουερθ. Συμφωνώ με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ότι είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η συμφωνία και πρέπει να στηριχθεί από την Επιτροπή σας. Σίγουρα δεν ήταν εύκολη η συμφωνία αυτή αν και υπάρχει η συμφωνία αυτή για την απελευθέρωση του εμπορίου στο πλαίσιο του ΕΟΧ, αλλά γενικώ ε, υπήρχαν κάποια ζητήματα που δεν είχαν ε, τεθεί σε διαπραγματεύσεις. Η Νορβηγία ξέρουμε ότι έχει έναν αρκετά μη παραγωγικό γεωργικό τομέα, πολύ υψηλή προστασία στα σύνορα, περιορισμένες δυνατότητες εξαγωγών και μεγάλο έλλειμμα διεθνούς εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Γι' αυτό και δεν ήταν τόσο πρόθυμοι για τις διαπραγματεύσεις αυτές ε, να συνεχιστούν δηλαδή. Βλέπουμε όμως ότι τελικά έγινε διαπραγματεύσεις βάσει των διατάξεων του ΕΟΧ και έχετε την πρόταση αναχείρας. Όπως σημειώνει και ο εισηγητής, ήδη έχει ε, υπάρξει περαιτέρω απελευθέρωση κατά 20% των εισαγωγών, άρα 60% ε, των εισαγωγών ε, είναι αδοσμολόγητες και υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε αρκετά διαχειρίσιμες ποσοστώσεις και μάλλον δασμούς. Τώρα, ποσοστός. ό,τι αφορά τα πορτοκάλια, Κάναμε το σχετικό αίτημα στις διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχει ένας τομέας ε, για τον οποίο η Νορβηγία ε, αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή της και είναι ο συγκεκριμένος τομέας αυτός. Οπότε ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε κάποια εξέλιξη με τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα πρόσφερε στις διαπραγματεύσεις αυτές ε, συγκρίσιμα αμοιβαία ανοίγματα για τις εξαγωγές, ε, τις νορβηγικές, αλλά επειδή όπως είπα είναι πολύ μικρό το δυναμικό εξαγωγής από την Νορβηγία, δεν περιμένουμε να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις των εξαγωγών της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε την έγκριση της συμφωνίας από το Νορβηγικό Κοινοβούλιο εντός Φεβρουαρίου και μετά από αυτό η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα υπογράψουν την ε, συμφωνία, ελπίζοντας βέβαια ότι υπάρχει και συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μετά θα τεθεί σε ισχύ βέβαια αυτή η συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Διευθυντή Κλάρκ και αν συμφωνεί και ο εισηγητής θα σταματήσουμε εδώ ε, υπενθυμίζοντα ότι θα πρέπει μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι να έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες και ότι θα, θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας την 7η ε, Φεβρουαρίου. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 12 λοιπόν της ημερησίας διατάξεως συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα. Ε, ξεκινάμε λοιπόν σε μια νομοθετικού περιεχομένου πρόταση πάρα πολύ σημαντική με μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η παρουσίασε τον προηγούμενο Δεκέμβρη την δέσμη για την ποιότητα ε, μετά από μια εκτενή δημόσια διαβούλευση ε, που ακολούθησε την δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για την ποιότητα το 2009. Ε, η Δέσμη προτείνει δύο προτάσεις κανονισμού καθώς επίσης και δύο κατευθυντήρες γραμμές. Ένα για τα συστήματα τυποποίησης και ένα για τις ετικέτες των προϊόντων που περιέχουν συστατικά PDO και PGI. Οι προτάσεις είναι πολύ εξαντλητικές και περιέχουν μερικά από τα σημεία τα οποία έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας ε, του συναδέρφου Γιανκάρλου Σκοτά. Επίσης ε, θα ήθελα να σας πω ότι ε, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα στοιχεία τα οποία αφορούν πράξεις νομοθετικές και κατεξουσιοδότηση που, και, που θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσουμε την εναρμόνιση τα επόμενα χρόνια. σήμερα θα, έχει, θα λάβει χώρα χώρα η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εμείς θα συνεχίσουμε την ε, συζήτησή μας σε, μια, ε, σε ένα εργαστήριο ad hoc, το οποίο θα λάβει χώρα τον, την 15η Μαρτίου 2011. Θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκπροσωπείται από την κυρία Μαρία Άγχελες Μπενίτε Σάλλας, που είναι διευθύντρια υπεύθυνη για την πολιτική ποιότητα της Γενικής Διεύθυνση Γεωργίας και μετά θα δώσουμε το λόγο στη δικιά μας συγγήτρια, κυρία Ιρέτκε Γκαρσία Πέρες. Μενείτε άλλες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια έστω και σύντομη παρουσίαση των προτάσεων αυτών ε, για την ποιότητα. Ένα πακέτο που όπως έχει πει πολλές φορές ο Επιτρόπος Τσεόλος ε, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της κοινή γεωργικής πολιτικής και αφού είναι ακριβώς ουσιώδες στοιχείο της ΚΑΠΑ Αυτά τα συστήματα έχουν, όπως ξέρετε, ε, αποτελέσει αντικείμενο μακρών διαβουλεύσεων και ε, ε, ανταλλαγής απόψεων σε μένους τομείς. Το 2008 είχαμε υποβάλει μια πράσινη βίβλο για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Συλλέξαμε απόψεις από χώρες, φορείς, ε, ενδιαφερόμενους. Το 2009 παρουσιάσαμε την ανακοίνωση που λάμπανε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις αυτές και έδινε κάποιου προσανατολισμούς που θα ήταν υπό μελέτη. Δεν θέλω να φάνονταν αποφάσεις στο επίπεδο της Κομισιόν. Και καρπός όλης αυτής της διαδικασίας είναι οι προτάσεις που μόλις υποβάλλουμε πριν από πολύ λίγες εβδομάδες. Και περιμένουμε να έχουμε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για την περαιτέρω επεξεργασία του. Το πακέτο ποιότητα, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, αποτελείται από δύο νομοθετικές προτάσεις. Η μία αφορά τα πρότυπα εμπορία και η δεύτερη αυτό που εμείς που καλούμε συστήματα ποιότητα, δηλαδή γεωγραφικέ ενδείξει ε, ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες και Πρόκειται και για δύο κείμενα συστάσεων που έχει ήδη αποφασίσει η Επιτροπή και μπορούν οι φορείς πλέον να τα χρησιμοποιούν. Το ένα φορά τη χρήση συστατικών υπογεωγραφική ένδειξη στα τρόφιμα και δεύτερο κείμενο σύστημα εθελούσιας πιστοποίησης. Ο στόχος μας με όλα αυτά είναι να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας να προβάλλουν και να αξιοποιήσουν περισσότερο και τα προϊόντα τους που συνδέονται συγκεκριμένα με μια περιοχή, με ένα έδαφος, το τερουάρο όπως λέμε, που αποτελεί παράδοση σε ό,τι αφορά τεχνογνωσία και να προβάλλουν επίσης και τα προϊόντα που έχουν μια ιδιαίτερη ιδιότητα ε, που θέλει να την κοινοποιήσει προς το καταναλωτή ο παραγωγός. Ό,τι αφορά την νομοθετική πρόταση. Και αναφέρομαι αρχικά στα πρότυπα εμπορίας. Το βασικό περιεχόμενο πέραν της προσαρμογής στους νέους κανόνες της συνθήκης της Λισαβόνας που είπατε κι εσείς ότι λαμβάνονται υπόψη εισάγει βασικό πρότυπο εμπορίας, που δεν νομίζω ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, γιατί αυτό που όλοι θέλουμε, όλοι οι καταναλωτέ θέλουν, είναι να είναι υγιεινό το προϊόν, να μπορεί να τεθεί στο εμπόριο. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα γενικό πλαίσιο, ώστε στο μέλλον να είναι δυνατό αν χρειαστεί να δημιουργηθούν και άλλα πρότυπα εμπορία πιο συγκεκριμένα, πιο ειδικά και βέβαια για να είναι δυνατόν αν εάν αυτό χρειαστεί και μετά βέβαια από ανάλυση μελέτη επιπτώσεων πιο αναλυτική ή ετικετοθεσία ε, προέλευση, το σήμα προέλευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το συζητήσαμε και στο θέμα της ενημέρωσης των ε, καταναλωτών που συζητείται στη, ε, στο πλαίσιο της συναπόφασης αυτή τη στιγμή και με το Κοινοβούλιο. Η πρόταση για την ποιότητα τώρα, δηλαδή για τα συστήματα ποιότητα συγκεκριμένα, στόχος αυτής της πρότασης είναι να διευκρινίσει και να πλουστεύσει ακριβώς αυτά τα συστήματα ποιότητας τα οποία υπάρχουν, είναι ήδη φυστάμενα ε, γεωγραφικές ενδείξεις, ονομασίες ε, προέλευσης, άλλα εγγυημένα συστατικά χαρακτηριστικά, δίνοντας μια νέα δυνατότητα κοινοποίησης συγκεκριμένων ιδιωτήτων. Προαιρετική όρη ποιότητας, έτσι το λέμε εμείς. Στόχος μας είναι τώρα να ορίσουμε καλύτερα το πεδίο εφαρμογή, να δώσουμε σαφέστερους ορισμούς, να διευκρινίσουμε τις σχέσεις μεταξύ γεωγραφικής ένδειξης και σήματο, μάρκα, γιατί μιλάμε και για προστασία τη πνευματική ιδιοκτησία. Θέλουμε να προστατευτεί ε, μια ονομασία. Επίση, στόχο μα ήταν να διευκρινίσουμε ή να αναγνωρίσουμε, θα έλεγα καλύτερα, το ρόλο των ομάδων παραγωγών. Επίσης διευκρινίσαμε διατάξεις για τον έλεγχο τη χρήση αυτών των ονομασιών και τις θέσεις του στο εμπόριο και κυρίω απλουστεύσαμε και μειώσαμε πάρα πολύ και τις διαδικασίες γιατί υπήρχαν βραδίες, μακρές διαδικασίες. Τις περικόψαμε, τις συμπνήσαμε και είναι πιο εύκολη έτσι η διαδικασία και διευκολύνεται και η ζωή όλων όσων χρησιμοποιούν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα συστήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ιδιαιτερότητες πλέον που εγγυόμαστε, που είναι εγγυημένες, ήταν πάρα πολύ πολύ το μέχρι τότε υφιστάμενο σύστημα και μάλιστα Ακόμα και εμείς στην Επιτροπή δυσκολευόμαστε να ερμηνεύσουμε κάποιες από αυτές τις ιδιαιτερότητες. Θέλησαμε λοιπόν αυτό το σύστημα να το περιορίσουμε στις ονομασίες εκείνες ή μάλλον στις εφαρμογές και υποψηφιότητες εκείνες που θέλουν, που ανταποκρίνονται σε κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και κυρίως για προϊόντα αναπτυγμένα ε, που έχουν παρασκευαστεί. Η γεωγραφική ένδειξη έχει σχέση με, τη σχέση με το έδαφος, το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι η τεχνογνωσία. Και προτείνουμε και ένα γενικό πλαίσιο που έχει προσθεθεί, ώστε να μπορούν να κοινοποιούνται κάποια συγκεκριμένα ε, χαρακτηριστικά ε, θελοντικής ε, αναφοράς, προαιρετικής δηλαδή αναφοράς. Το πακέτο αυτό συμπληρώνεται, όπως είπα και στην αρχή, με δύο ανακοινώσεις της Κομισιόν, με κατευθύνσεις γενικές πρώτων σε ό,τι αφορά τα συστατικά. Συγγνώμη, για να το ξαναπώ. Συστατικά βάσο, ε, υπογεωγραφική ένδειξη που χρησιμοποιείται σε άλλα τρόφιμα. Κατά την απόψή μου. Συστάσεις κοινού νου θα τις έλεγα κοινή λογική, ώστε να ενημερωθεί καλύτερα ο καταναλωτή για αυτέ τι γεωγραφικέ ενδείξει. Και επίση υπάρχει και μια σειρά κατευθύνσεων για τα συστήματα θελούσια πιστοποίηση που στόχο έχουν να ενισχύσουν τη θέση των παραγωγών στι διαπραγματεύσει αυτέ και να του δώσουν τη δυνατότητα να έχουν όλα τα όπλα που μπορούν να διαθέτουν για να προσπίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να την προβάλλουν. Ε, κατά κλείδι, κυρίες και κύριοι, με αυτό το πακέτο, ο στόχος μας είναι να δώσουμε ένα γήπεδο ε, στο οποίο θα μπορούν να παίξουν οι παραγωγοί, να μπορούν να ενημερώσουν καλύτερα τους καταναλωτές, να προβάλλουν καλύτερα τα προϊόντα τους και να έχουν και μια πιο δίκαια τιμή για τα προϊόντα που προσφέρουν. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με πολύ μεγαλύτερε λεπτομέρειες και μαζί σας ε, τους επόμενους μήνες ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία της συναπόφασης που βρίσκεται στη συνήθιδη, εντάξει, την κανονική διαδικασία στο επίπεδο της Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την ε, κυρία Μπενίτε Σάλλας και θα δώσουμε τώρα τον λόγο στη δικιά μας εισηγήτρια. Η Ράτσα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς βέβαια να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίαση που έκανε. Εμείς είμαστε βέβαιοι στην Επιτροπή μας ότι υπάρχει συμφωνία σε ό,τι αφορά το ότι η ποιότητα των γεωργοδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων είναι η ταυτότητα ε, της ε, γεωργίας μας. Είναι ένα σημαντικός παράγοντας για να στηρίξουμε και την ανταγωνιστικότητα του τομέα και βέβαια να ανταποκριθούμε και στους καταναλωτές οι οποίοι ζητούν παραδοσιακά προϊόντα τα οποία αναπτύσσονται με συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής. Έχω κάποια πολύ σύντομα ε, ζητήματα που θέλω να θέσω και θα δώσω μετά το λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Θεωρώ πάρα πολύ θετική τη διατήρηση των τριών συστημάτων για τις διάφορες ονομασίες. Και εμείς ε, είχαμε πει ότι πρέπει ιδίω να παραμείνει η τρίτη συγκεκριμένα κατηγορία που αφορά τις ιδιαιτερότητες και για το PDO, για το παραδοσιακό χαρακτήρα δηλαδή ενός προϊόντος, ε, πρέπει να έχουμε την κατάλληλη προθεσμία. Θα ήθελα να ακούσω όμως και άλλους ε, συναδέλφους τι έχουν να πούν. Η Ευρωπαϊκή Πετροπή Προσπαθεί να βελτιώσει και να απλουστεύσει ε, τα δύο συστήματα, τα γεωγραφικά, δίνοντα ένα υψηλό επίπεδο προστασία που θα πρέπει να μετωσιωθεί και εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη. Με βάση τα συστήματα ποιότητα, γεωγραφικέ ενδείξει και ονομασίε προέλευση να είναι κοινέ, γνωστέ στην κοινή γνώμη. Πώς βλέπετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Στρέφομαι να υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να δώσουν εργαλεία σε ομάδες παραγωγών οι οποίοι στους οποίους προσωπούνται όλοι οι φορείς της αλυσίδας της παραγωγής αγορο, ε, των προϊόντων. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ο κλάδος δεν έχει ακόμη εισακουστεί στις ανησυχίες που έχει τη δυνατότητα εκχώρησης κάποιων αρμοδιοτήτων σε ομάδες αυτές ε, παραγωγών. Ένα άλλο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, συμφωνία της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο, όταν δηλαδή εγκρίναμε την έκθεση Σκότα για τα θέματα αυτά. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε γιατί έχει εξαφανιστεί το προϊόν ε, ορεινής γεωργίας στην τελική πρόταση την οποία μας υπέβαλε η Επιτροπή. Τώρα, για αυτούς τους προαιρετικούς όρους ποιότητας ε, και σε σχέση με, την, ε, με τους όρους εμπορίας. Ε, γιατί διαχωρίζεται αυτό από τον κανονισμό για την ενιαία ΚΟΑ. Στον κανονισμό ποιότητας επίσης, επίσης διαχωρίζονται από τα στοιχεία τα οποία αφορούν τα στοιχεία της ποιότητας. Ό,τι αφορά τώρα προτινόμενες αλλαγές στην ενιαία ΚΟΑ με βάση τα πρότυπα εμπορίας, είναι πιο τεχνικές οι πτυχές και νομίζω πρέπει να μπορέσουμε να τις εξετάσουμε αναλυτικά. Υπάρχουν αρκετές διατάξεις οι οποίες θα αναπτυχθούν μέσω εξουσιοδότηση πράξεων. Ως εισηγήτρια στόχο έχω να επιδιώξω την εξισορρόπηση μεταξύ της τεχνικής ταχύτητας της Κομισιόν για να αναπτύξει αυτές τις διατάξεις και των βασικών σημείων από τον οποίο αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρήσει το ρόλο του συνομοθέτη. Και δύο πολύ συγκεκριμένα θέματα. Η πρόταση περιλαμβάνει τα παραρτήματα του υφιστάμενου κανονισμού που 1204-2007 ό,τι αφορά όμως ε, το κρέας ε, και τα πτηνά υπάρχουν κάποια πολύ ουσιαστικά σημεία των προτύπων τα οποία έχουν διαγραφεί και σε ό,τι αφορά ε, τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ειδικά όρου ποιότητα. Ε, Γι' αυτό τα προϊόντα θα ισχύουν ε, τα γενικά πρότυπα των οργανισμών εναρμόνισης. Τι συμβαίνει με ένα σύστημα πιστοποίησης ταξινόμησης που λειτουργεί ήδη καλά σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι νομίζω θέματα γενικά στα οποία θα ήθελα να έχω κάποιε απαντήσει, να ακούσω τη θέση τη Κομισιόν, να έχω κάποιε εξηγήσει. και όπω είπα αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων, των σκιωδών από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Στόχος μου είναι να συνεργαστώ με όλη την Επιτροπή, με όλα τα μέλη της Επιτροπής, ώστε να καταλήξουμε σε μία ώστε να τον πιο ομόφωνη θέση του Κοινοβουλίου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη όλες μας τις ανησυχίες και όλες μας τις απόψεις, ώστε να μπορέσουμε και στη συνέχεια να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο ένα πακέτο το οποίο θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες όλων. Ευχαριστούμε πολύ Ράτσε. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Θα ήθελα όμως να μην ξεχνάτε τις σημαντικές ημερομηνίες. 15 Μαΐου 2011 ειδικό εργαστήριο για την ποιότητα. 28 ε, Μαρτίου ε, συζήτηση του σχεδίου έκθεσης. 11 ε, Απριλίου 2011 η προθεσμία για την υποπολή τροπολογιών και 25 Μαΐου 2011 η έγκριση ψηφοφορία και ενδεχομένω έγκριση. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τους συναδέλφους, πρώτα απ' όλα η Σέλφος Ρέιμερς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν ε, χαίρομαι διότι υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί οι οποίοι θα συγχωνευτούν γιατί η ποιότητα είναι βασική για τα γεωργικά προϊόντα. Ζητάμε υψηλέ προδιαγραφές από τους γεωργούς μας αλλά πρέπει να μπορούμε να του συνδράμουμε στο θέμα του μάρκετινγκ και επίσης θα ήθελα αυτό να καταστεί υποχρεωτικό. Δηλαδή ε, έτσι θα υπάρχει και ένα επιπλέον ε, μέσο marketing διότι όταν ε, όλοι πρέπει να συμμετέχουν είναι κάτι που δεν αντιλαμβανόμαστε στο marketing και στη διαφήμιση. Για μένα θα ήταν μια υποχρεωτική διαδικασία διότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα αυτή. Και γι' αυτό θα θα ήθελα να προσθεθεί και αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Herbert Norfeld. Και εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται στην κατάλληλη στιγμή και ε, είναι μια εξαιρετική πρόταση. Είναι καλή πρόταση διότι πρέπει να ε, ε, ενοποιηθούν οι ονομασίες προελεύσεως και πιστεύω ότι είναι σωστό όσον αφορά το κρασί να το αφήσουμε εκτός όχι γιατί δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο για αυτό το προϊόν αλλά διότι έχει υπάρξει προσφάτως μια νέα ρύθμιση και χρειάζεται να επέμβουμε και πάλι τώρα. Όσον αφορά την ε, ονομασία προελεύσεως, βλέπουμε ότι σε πολλά κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Γαλλία υπάρχει μία μεγάλη ε, παράδοση ενώ στη Βόρειο Ευρώπη δεν είναι ίδια η κατάσταση. Άρα η πρόταση η οποία ε, προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ε, μπορέσει ε, να ρυθμίσει αυτά τα θέματα, να προσφέρει μία επιπρόσθετη προστασία διεθνώς και θα μπορεί να τα προστατεύσει τα προϊόντα και εντός της Ευρώπης. Παραδείγματος χάρη αναφέρομαι στην Παρμεζάνα ή σε την πύρα Είναι θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και εντός της Ευρώπης. Τώρα, ε, ήδη ανέφερε η συγγήτρια ότι ένα βασικό θέμα συζήτηση είναι ο ρόλος των χριστών. διότι είναι προφανές ότι οι συνάδελφοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπαν σήμερα ότι ε, οι ονομασίες προελεύσεως είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες για όλους αλλά οι ορισμένες ονομασίες προελεύσεως παίζουν ρόλο μίας μάρκας και πρέπει να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τα δύο στοιχεία. Δηλαδή ο χρήστης θα μπορεί να επηρεάζει περισσότερο τη διαμόρφωση ε, αυτής της προβολής, δηλαδή ε, να υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση ε, στην χρήση αυτών των ονομασιών προελεύσεως, γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ευρώπη όπου δεν υπάρχει μία μία συντονισμένη κίνηση από πλευράς εμπορίας και προωθήσεως και δεν έχουν επιτευχθεί ε, οι αναγκαίες ε, επιτυχίες. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε και να προσέξουμε επίσης την επεξεργασία των προϊόντων διότι αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και ενδεχομένως θα μπορούσα να αναφέρω σαν παράδειγμα ότι αν μιλάμε για προσούτο διπάρμα τότε εάν μιλάμε για ένα σάντουιτς είμαι πολύ επιφυλακτικός. Οπότε θα πρέπει παραδείγματο χάρη ε, να ε, ε, είναι ελέγξιμα τα στοιχεία. Επίσης όταν μιλάμε για προϊόντα ορεινών περιοχών ε, όταν θα αριθμιστεί αυτό το θέμα διότι γνωρίζω ότι η πρόταση αυτή ε, υπήρχε και περιλαμβανόταν στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την τελευταία στιγμή εξαφανίστηκε για άγνωστους για μένα και ακατανόητους λόγους. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να περιληφθεί διότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι ορατά και για τους καταναλωτές. Ο κύριος Ντοντέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο συνάδελφος Σκότα παρουσίασε μία έκθεση η οποία έγινε γενικά αποδεκτή από το Κοινοβούλιο και τώρα προσπαθούμε ε, μέσω τροπολογιών να επαναλάβουμε αυτά που ελέγονται στην έκθεσή του και δεν βρίσκουμε σε αυτήν θα ενισχύσουμε τα επιχειρήματά μας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις επαναφέροντας το θέμα της ονομασίας προελεύσεως στον ΠΟΕ. Αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να αναφέρω. Παραδείγματος χάρη το θέμα των προτάσεων για την προέλευση από ορεινές περιοχές που υπήρχε στην αρχή αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει πλέον και δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της απόσυρσης. Ξέρουμε ότι η έκθεση Σκότα τόνιζε σαφέστατα ότι υπάρχει ε, μία σύνδεση στην προστιθέμενη αξία μεταξύ της διαχείρισης ε, της ε, ονομασίας και διαχείρισης των όγκων των ποσοτήτων, πράγμα το οποίο δεν επανελήφθη στην έκθεση και εδώ Α αναφέρουμε στον κύριο Ντικάστρο γιατί πιστεύω ότι και οι δύο θέλουμε να επαναφέρουμε μέσω τροπολογιών αυτό το στοιχείο. Επίσης όσον αφορά τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν δεν κατάλαβα σχετικά με τα ε, STG που θα ε, περιοριστούν στα μεταποιημένα προϊόντα και δεν ε, θα υπάρξει σε αυτή την ονομασία και σε αυτό τον καθορισμό για ε, προϊόντα τα οποία καταρχήν είχαν προβλεφθεί αλλά τώρα εγκαταλείφθηκαν. Ευχαριστώ. Πολύ σαφές. Τώρα θα προσθέσω και εγώ. Ε, αλλά στο τέλος και προς το παρόν θα δώσω λόγο στον κύριο Σμιτ. Θα είμαι σύντομος διότι ε, νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει στην επόμενη, στη σωστή κατεύθυνση διότι πολλοί από εμά συνέβαλαν στη διατύπωση αλλά καλό θα ήταν να παρουσιάσουμε την προστιθέμενη αξία και να μην αναφερόμαστε μόνο στο ότι υπάρχει ένα ειδικευμένο προϊόν με προστιθέμενη αξία και ε, όχι μία γενίκευση ε, στα γεωργικά προϊόντα. Υπάρχουν ε, εξειδικευμένες αγορές, niche markets και αυτά πρέπει να επιζητήσουμε. Ε, πρόκειται όμως για διαφορετικές ε, κινήσεις ε, στο ίδιο περιβάλλον και γι' αυτό χαιρετίζω αυτόν τον χαρακτηρισμό. Επίσης εγώ είμαι Σκοτσέζος και συμφωνώ ότι πρέπει να τονίσουμε την ορεινή προέλευση και να περιλάβουμε στις προελεύσεις γεύσεις πέραν των ωραίων αλλά και τα, ε, και τα νησιά διότι πιστεύω ότι όλα αυτά προσθέτουν αξία στα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σμίτ. Καλινόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θέλω να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Επιτροπή αποφάσισε τελικά να ε, κάνει τόσο μικρό κατάλογο προδοσιακών προϊόντων και γιατί αποφάσισε ε, να περιλάβει μονάχα επεξεργασμένα ε, προϊόντα. Εμεί θα προτιμούσαμε και τα μη επεξεργασμένα προϊόντα να συμπεριληφθούν, γιατί διαφορετικά το θέμα δεν γίνεται πολύ ελκυστικό για τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, δεν είναι καθόλου σαφές τι εννοούμε με το επεξεργασμένο προϊόν. Όλα τα, προγρα... όλα τα προϊόντα τα οποία είναι καταγραμμένα αυτή τη στιγμή στο σύστημα υποτίθεται ότι έπρεπε να καλυφθούν στο νέο σύστημα λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι ο κανονισμός θέτει νέα ε, στοιχεία, νέα κριτήρια για την καταγραφή. Δεν θα πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια πριν ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στην ε, Διευθύντρια κυρία Μπενίτες Σαλάσα. Υπογραμμίζω αυτά που είπε μόλις τώρα ο συνάδελφος Μισελ Νταντά. Υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία της έκθεσής μας, ε, έκθεση σκοτά για την ε, ποιότητα, που υπερψηφίσαμε εδώ στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, που ε, περιλαμβάνουν επιχειρηματολογία που όμως δεν έχει συμπεριληφθεί σε αυτήν την δέσμη για την πρόταση, κυρίως όσον αφορά ε, την τον παραγωγικό προγραμματισμό, θέμα του οποίου είχαμε εκφράσει σαφώς την άποψή μας. Επίσης, ε, ειδικά προϊόντα από ορεινές περιοχές κτλ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω, αν μου επιτρέπει, μια ερώτηση στην εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας. Για αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη πιστοποίηση βάσει της γεωγραφικής τους προέλευσης και που μέσα από την νέα νομοθετική πρόταση θα πρέπει να αλλάξουν όνομα ή τέλος πάντων να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις γιατί το όνομά τους δεν είχε καταγραφεί ας πούμε η ε, ε, ναπολιτάνικη πίτσα θα πρέπει να προβλεφθεί ε, ε, μία ε, μία διαδικασία προτιμησιακή γιατί διαφορετικά το 2017 βάσει αυτής της νέας δέσμης για την ποιότητα δεν θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να καταγράψουμε την Ναπολιτάνικη πίτσα ως προϊόν ειδικής γεωγραφικής προέλευσης. Προβλέπετε λοιπόν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά ξανά στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, βλέποντας την έκθεση Σκότα, νομίζω τα σημεία που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία λαμβάνει υπόψη της η Κομισιόν. Τα αποδέχεται. Άρα νομίζω από αυτήν την έννοια μπορεί να εκτιμηθεί θετικά η πρότασή μας. Τώρα, τα ζητήματα που αναφέρθηκαν επανειλημμένως. Ας ξεκινήσω όχι με το πιο εύκολο, γιατί η πρόταση αυτή είναι με πλή, αλλά δεν είναι εύκολη σε ό,τι αφορά κάποιες προαιρετικές ενδείξεις που αναφέρονται. Θέλαμε να τις ε, συμπεριλάβουμε ε, στον κανονισμό 1634, αλλά είχαν, ε, ήταν διάσπαρτες σε διάφορους τομεακούς κανονισμούς. Θέλαμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να τα συνενώσουμε και να τα καταστήσουμε συνεκτικά και νομίζω ότι αυτό είναι ήδη μια σημαντική συμβολή. Στόχος μας δεν είναι να εξαρθρώσουμε αυτό το οποίο υπάρχει ήδη, ανέφερε η συγγήτρια. Ε, τα αυγά και το κρέας των πτηνών. Αυτό δεν εξαφανίζεται από το κείμενο. Υπάρχει μια μεταβατική διάταξη που επιτρέπει να μεταβούμε από τους υφιστάμενους κανόνες σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Ξεκολουθούν λοιπόν όλα να ισχύουν μέχρι ότου εγκριθεί από την Κομισιόν ή αραντίστοιχη κάθε φορά κατεξουσιοδότηση πράξη. Σε ό,τι αφορά τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο ανέφεραν περισσότεροι βουλευτές, τι ορεινέ περιοχέ, γιατί δεν υπάρχει πλέον στην πρότασή μα, γιατί εξαφανίστηκε η πρόταση που είχε μελετηθεί για τι ετικέτε των ορεινών προϊόντων. Να σα πω γιατί. Είναι περίπλοκο το ζήτημα και θέλουμε τι αναλύσεις, τι εσωτερικέ αναλύσεις και τη συλλογή δεδομένων, θέλουμε να την ολοκληρώσουμε κατά τρόπο ώστε να μπορούμε να προτείνουμε ένα πρότυπο, έναν κανόνα που θα είναι ω το δυνατόν πιο συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο σε διαφορετικέ πραγματικότητε ώστε να τον πιο κοντά στι διαφορετικέ πραγματικότητε, ώστε να είναι χρήσιμο προ του ε, χρήστε. Να μην είμαστε μόνο στα όρια γενικόλογων ε, διατάξεων. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε πραγματικά μεγάλη ε, κατακραυγή θα έλεγα και υπήρχε τέλος πάντων αντίδραση. Αλλά θέλαμε εμείς να έχουμε μια πιο προσαρμοσμένη πρόταση σε ό,τι αφορά αυτά τα εγγυημένα ε, χαρακτηριστικά. Ο, ίδιος ο που ήδη ισχύει είναι λίγο πολύπλοκος. Μιλάμε για ένα σύστημα ετικετοθεσίας, όχι για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις ετικέτες ξεκολουθεί να προβλέπεται η δυνατότητα να γραφεί ένα προϊόν με ή χωρίς ε, επιφύλαξη ονομασίας. Δηλαδή υπάρχουν κάποια προϊόντα που μπορούν να εξακολουθήσουν να ονομάζονται με τον ίδιο τρόπο και να κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ποιο, ε, ποια είναι τα ε, πλεονεκτήματα για τον παραγωγό και ποια είναι η σαφήνεια και πώ ε, εννοεί τα πράγματα ο καταναλωτής. Θα ήθελα να διαβάσετε, γιατί είναι στο σελίδα μα η μελέτη επιπτώσεων που δίνει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που θα σα διαφωτίσουν. Ένα σύστημα λοιπόν πολύ πιο σαφέ ω προ τη σύλληψή του θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εποφελές για τον παραγωγό και πολύ πιο σαφέ για τον καταναλωτή και συγκεκριμένα για τα καταχωρισμένα είδη προϊόντα. Θελήσαμε να υπάρχει ένα μεταβατικό σύστημα κανόν, θα το συστήσουμε μαζί σα, ώστε να μην πληγούν σε καμία περίπτωση τα είδη καταχωρισμένα προϊόντα. Για κάποια βέβαια υπήρξε ε, και κάποιο όφελο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα άλλο θέμα που ανέφεραν πολύ για τους παραγωγούς συγκεκριμένα. Η πρόταση αυτή τη στιγμή αναγνωρίζει ρητός το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι όμιλοι παραγωγών, οι ομάδες παραγωγών, σε ό,τι αφορά το συντονισμό τους, ε, των παραγωγών δηλαδή, την ενημέρωσή τους, ε, οικονομικές γνώσεις, ε, παρακολούθηση και της παραγωγής, των ιδιαιτεροτήτων, των όρων της αγοράς κτλ. Αυτό τώρα που έχει να κάνει με τη διαχείριση όγκων μας φαίνεται λίγο πιο προβληματικό. Γιατί δεν μπορεί να προβλεφθεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ένας γενικός κανόνας, ένα γενικό πρότυπο από αυτήν την έννοια γιατί αυτό πιστεύουμε ότι θα αφορούσε πολύ άμεσα και ίσως θα ερχόταν και σε αντίθεση με τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Έτσι ώστε ό,τι έχει να κάνει με διαχείριση όγκων. Παίρνω το ότι εμεί θεωρούμε ότι ήδη το κοινοτικό δίκαιο παρέχει κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες και πρότυπα που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το γάλα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λοιπόν. Επομένω, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, να μελετούμε δηλαδή τη διαχείριση των νόμων, αυτό θα πρέπει να γίνει κατά περίπτωση και όταν το δικαιολογούν οι συνθήκες. Δεν ανοίγω κανένα παραθυράκι κύριε Πρόεδρε, έτσι σε καμία περίπτωση. Απλά σας μίλησα για το παράδειγμα της δέσμης μέτρων για το γάλα. Είπα ότι πρέπει να το μελετήσουμε σε πολύ μεγαλύτερο βάθος για να δούμε τι σχέση υπάρχει με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ελευθερία των παραγωγών να παράγουν τα προϊόντα τους και την επιλογή των καταναλωτών, το δικαίωμά να επιλέγουν. Και αυτά διείπαν και τις προτάσεις που έχετε αναχείρες. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η Ράτσε θέλει να πει δύο λόγια πριν ολοκληρώσουμε. Η Ράτσε, Γερσία Πέρες, έχει το λόγο. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις απαντήσεις που έδωσε. Υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και για κάποια άλλα. Καλό θα ήταν ίσως να γίνει μια προσπάθεια διαλόγου και κατανόησης ή συνεννόησης αν θέλετε. Ε, οι περισσότεροι συνάδελφοι έθεσαν κάποια θέματα τα οποία εμείς, για τα οποία εμείς τοποθετηθήκαμε μέσω της έκθεσης Σκότα. Τη στηρίζει δε αυτές τις προτάσεις και η πλειοψηφία των βουλευτών. Είμαι πεπισμένη ότι ο στόχος τόσο της ε, Επιτροπής όσο και του Κοινοβουλίου είναι ο ίδιος, δηλαδή να βελτιώσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Επομένως, επόμενους μήνες θα έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε. Παναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου προς τους βουλευτές που έλαβαν τον λόγο και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μέσα το δυνατόν πιο συνενετική κοινή πρόταση. Άψογα να σας υποθυμίσω ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι 15 Μαρτίου, workshop για την ποιότητα, ε, συζήτηση του προσχεδίου έκθεσης 28 Μαρτίου, 11 Απριλίου η προθεσμία υποβολής τροπολογιών, ψηφοφορία στην Επιτροπή 25 Μαΐου. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Υπενθυμίζω ότι ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις με τους συντονιστές. Έχουμε ορίσει λοιπόν αρκετές εκθέσεις πρωτοβουλίες. Καλό είναι να έρθει σε επαφή με τους συντονιστές της κάθε ομάδας, ο καθένας με την ομάδα του. Υπενθυμίζω ότι στις 3 το απόγευμα θα ξεκινήσουμε την μεγάλη ακρόαση για την κοινή γεωργική πολιτική στην Ολομέλεια, στην έψο της Ολομελίας. Ε, καλό μεσημέρι, καλή όρεξη. Oui, le 2. Exactement.